Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να φάγατε καλά. Εγώ τουλάχιστον έφαγα καλά το μεσημέρι. Πρέπει να πω ότι μέχρι τώρα δεν είμαστε εδώ πολλοί, αλλά να ήδη βλέπω έναν από τους δύο συνεισηγητές που μπήκε στην αίθουσα και κάθεται. Ωραία, οπότε χαίρομαι που μπορώ να σας καλωσορίσω όλους σε αυτήν την κοινή συνεδρίαση που έχουμε με την Επιτροπή Στεγματικών Υποθέσεων. Για νομικούς λόγους μου είπαν ότι πρέπει να σας ενημερώσω ότι η συνεδρίαση αυτή θα αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο. Όποιος δεν έχει τη συνήθεια και δεν θέλει να αναμεταδοθεί από το διαδίκτυο ότι πει θα πρέπει να καταλήψει την αίθουσα. Λοιπόν, η μερίσια διάταξη. Εγκρίνεται, έχετε, έχει κυκλοφορήσει αν ε, δεν θέλετε καμία τροποποίηση, τότε θεωρείται εγκεκριμένη μερίσια διάταξη. Καλώς. Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση, η κοινή των Επιτροπών Συνταγματικών Υποθέσεων και Αναφορών όσον αφορά την ε, έρευνα της Ombudsman σχετικά με την ε, διαφάνεια στις συζητήσεις νομοθετικού περιεχομένου στις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συγητές είναι ο κύριος Λάινεν και η κυρία Τόμ που στις 13 Σεπτεμβρίου σας ε, έστειλαν το σχέδιο έκθεσης. Τα πρακτικά τα έχετε δει, θεωρούνται εγκεκριμένα, συμφωνείτε, της προηγούμενης ε, συνεδρίασης, ναι. Δεν θέλετε καμιά τροποποίηση, τίποτα. Ωραία, εγκρίνονται. Σημείο 4 τώρα λοιπόν, που είναι και η έρευνα της Ombudsman όσον αφορά τη διαφάνεια στη συζήτηση νομοθετικού περιεχομένου στις προπαρασκευαστικές ε, συζητήσεις των σωμάτων του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσω πρώτα το λόγο πέντε λεπτά στον καθένα από τους δύο εισηγητέ. Η κυρία Τουμ όμως πρέπει να σας πω ότι είπε ότι θα καθυστερήσει γιατί η πτήση, η πτήση της καθυστερεί. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι εδώ πριν το τέλος αυτής της συνάντησης. Όταν αφιχθεί, θα της δώσουμε και το λόγο. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας για αυτή την κοινή συνεδρίαση επιτροπών είναι λίγος. Κύριε Λάινεν, θα σας δώσω το λόγο που είσαστε συνεισηγητής εκ μέρου της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Για πέντε λεπτά έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Συμπρόεδρε. Πράγματι, Έχουμε μια πολύ σημαντική υπόθεση εδώ, ένα σημαντικό φάκελο. Πώς δηλαδή να ανοίξουμε αυτό το μαύρο κουτί των ενός εκ των διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Συμβουλίου. Η Ombudsman σωστά καταδεικνύει κάποιες από τις αδυναμίες που έχουν να κάνουν με την έλλειψη ακριβώς διαφάνειας στο Συμβούλιο. δεν πρόκειται για ένα διοικητικό σώμα, πρόκειται για ένα νομοθετικό ε, σώμα, όπως είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεπώς και οι δύο συνεισηγητές θέλουμε να υποβάλουμε μια πολιτική έκθεση και όχι μια τεχνική έκθεση. Είναι ιδιαίτερα πολιτική έκθεσή μας λοιπόν και θίγει κυρίως την ανισορροπία που υπάρχει όσον αφορά την διαφάνεια και την ε, προσβασιμότητα μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη μια, που επεξεργάζεται με απόλυτη διαφάνεια ε, τα πάντα στη νομοθετική διαδικασία και από την άλλη μεριά το Συμβούλιο, που όπως σας είπα είναι κάπως ένα κλειστό κουτί. Θέλουμε λοιπόν να ζητήσουμε από τους συναδέρφους και των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών, αλλά και τους υπόλοιπους, να επικεντρωθούν στο πεδίο εφαρμογή τη έκθεση αυτή και να μην υποβάλουν τροπολογίε οι οποίε να έχουν να κάνουν με όλα τα ζητήματα διαφάνεια ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Υπάρχουν ε, διάφορε εκθέσει που είχαμε κατά το παρελθόν με αυτό το σκοπό. Και υπάρχουν άλλε ευκαιρίε όπου θα μπορούσε κανεί να θίξει τέτοια ζητήματα γενικότερα διαφάνεια. Τώρα, κυρία πτυχή τη ε, έκθεση αυτή, ποια είναι. Στα συμπεράσματά μας λέμε ότι η τήρηση των συστάσεων της Ombudsman είναι το ελάχιστο προκειμένου να καταστεί περισσότερο διαφανής η νομοθετική διαδικασία στο Συμβούλιο. Θα μπορούσαν να γίνουν παραπάνω πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν διαφάνεια στην νομοθετική διαδικασία. Είναι αναγκαία για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να υποστηρίξει και να ενισχύσει την διαφάνεια αυτή. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται και η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Οι πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης και όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητούν από τους εκλεγμένους τους να λογοδοτούν. Χρειάζεται υψηλός βαθμός διαφάνειας λοιπόν, γιατί αποτελεί ρήτρα ασφάλειας κατά των fake news, των ε, υπερβολών Πιστεύουμε επίσης ότι η έλλειψη διαφάνειας στο Συμβούλιο έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν οι πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, οι ενδιαφερόμενοι, να μην μπορούν να ελέγξουν την συμπεριφορά των κυβερνήσεών τους. Επίσης εμποδίζει τα εθνικά κοινοβούλια να ελέγχουν τις ε, δράσεις των κυβερνήσεών τους στο Συμβούλιο και οδηγεί και σαν ισορροπία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επικρίνουμε επίσης το γεγονός ότι το Συμβούλιο πολύ συχνά αποφασίζει χωρίς να ψηφίζει. Ακόμα και για πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αποφασιστούν με ειδική πλειοψηφία. Το γεγονό ότι δεν γίνεται ψηφοφορία στο Συμβούλιο έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δούμε τελικά ποιο ψήφισε τι. Ποιο ήταν υπέρ, ποια κυβέρνηση ήταν υπέρ και ποια ήταν κατά μια απόφαση. Δεν μπορεί κανείς έτσι να γνωρίζει τη θέση της κάθε κυβέρνησης. Στη δημοκρατία όμως είναι λογικό να είσαι μερικές φορές στην πλειοψηφία, μερικές φορές να είσαι στην μειοψηφία. Διαφάνεια όμως πρέπει να υπάρχει για το τι ψηφίζεις, ό,τι και αν είναι αυτό. Έτσι λοιπόν ζητάμε από το Συμβούλιο να πάει ακόμα πιο πέρα και από την τήρηση των ε, συστάσεων της Ομπουτσμαν και να φροντίσει στις συνεδριάσεις της Κόρεπερ να υπάρχει αναμετάδοση στο διαδίκτυο. Να υπάρχει πρόσβαση δηλαδή από το κοινό, όπως γίνεται εδώ σε αυτή την ε, συνεδρίαση, αλλά και στις άλλες συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου που γίνεται αναμετάδοση στο διαδίκτυο έφτασε η στιγμή το Συμβούλιο να πάψει να λειτουργεί σαν ένα διπλωματικό φόρουμ και να αρχίσει να λειτουργεί σαν ένα νομοθετικό σώμα σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τέλος, προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα για το Eurogroup στην έκθεσή μας. Είναι μια βαστική ομάδα στο Συμβούλιο και νομίζω ότι πρέπει να τυποποιηθεί, για την άτυπη τώρα και θα έπρεπε οι κανόνες να ισχύουν και εκεί. Προσβλέπω στις παρατηρήσεις σας ε, τώρα και στα σχόλιά σας. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως, μας διαφωτίσατε και για μερικούς ήταν μια πολύ διαφωτιστική επανάληψη. Ωραία, είπαμε ότι για να το δεν είναι εδώ, μόλις φτάσει θα της δώσουμε το λόγο. Οπότε τώρα, εγώ έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω εγώ. Θα δώσω το λόγο στην Συνπρόεδρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Στο όνομα της ΑΦΚΟ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είχαμε δύο συναντήσεις πριν το καλοκαίρι με την Ευρωπαία Μεσολαβήτρια. Η μία ήταν κοινή συνάντηση μαζί σας και συζητήσαμε την έκθεση αυτή προτού να είναι διαθέσιμα τα σχετικά συμπεράσματα. Και κατόπιν είχαμε κοινή συζήτηση για τα συμπεράσματα της ε, στρατηγικής έρευνας. Και νομίζω ότι σαφές συμπέρασμα ήταν ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε το ίδιο επίπεδο διαφάνειας σε όλα τα θεσμικά όργανα. Θέλουμε λοιπόν να θίξουμε το θέμα. Ήδη αναφέρετε κάποιες ε, διαφορές όσον αφορά και την ε, πολιτική ε, νοοτροπία. Δεν μιλάμε όμως μόνο για αυτήν, μιλάμε και για την νομοθετική διαδικασία, όπου υπάρχουν κάποιες πρόσθετες απαιτήσει διαφάνειας και λογοδοσίας. Θα ήθελα επίσης να πω λίγα λόγια σχετικά με το τι αποφασίσαμε τον Ιούλιο κατά την πρώτη συζήτηση αποφασίσαμε το Συμβούλιο να παρέχει πληροφορίες στο Κοινοβούλιο, στις επιτροπές του Κοινοβουλίου, σχετικά με το πώς σκοπεύει να βελτιώσει τους κανόνες και την διαδικασία όσον αφορά την νομοθετική διαφάνεια. Λυπούμαστε που δεν ε, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα σήμερα. Παρ' όλα αυτά, αν θέλει κάποιο να πάρει το λόγο από το Συμβούλιο, θα χαρούμε πολύ. Η Γιάννα δεν είναι παρούσα. Θα ξεκινήσουμε από του σκιώδει εισηγητέ. Ε, από πλευρά τη Επιτροπή ΠΕΤΗ, λοιπόν, έχουμε τον Πέτερ Γιάρ. Μήπω θα ήθελε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ που επιτέλους ε, φαίνεται να προχωρούν τα πράγματα. Ε, αυτό το οφείλουμε στη διαμεσολαβήτρια. Η διαφάνεια θα μπορούσε να πει κανείς ε, ότι είναι ένα σύγχρονο σύνθημα, αλλά όχι, μπορεί να ε, βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς πραγματοποιείται η νομοθετική διαδικασία. Το κοινοβούλιο μας είναι πάρα πολύ διαφανές. Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την, ε, το πώς ψηφίζει ο κάθε ε, ευρωβουλευτής, ενώ το Συμβούλιο είναι ένα μαύρο κουτί, black box. Και μπορεί κανείς να πει ό,τι θέλει για τον κανονισμό περί διαφάνειας. Ε, ήταν όμως σε μια κοινή απόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Πολλοί πολίτες στην Ευρώπη δεν θεωρούν πολύ καλά τα όσα γίνονται, διότι ε, νομίζουν ότι η Γερμανία δεν συμμετέχει καθόλου στην νομοθετική διαδικασία. Νομίζω όμως ότι με διαφάνεια ε, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερη επιχειρηματολογία. Συμφωνώ λοιπόν, η πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τι έχει ψηφίσει το κάθε κράτος μέλος, ενδεχομένως και γιατί. Συνήθως δεν πρόκειται για ε, ε, κοσμοϊστορικά γεγονότα στο κάτω-κάτω. Εμεί, οι ευρωβουλευτές ε, συχνά δεν γνωρίζουμε πώς έχουν ψηφίσει τα κράτη-μέλη μας στο Συμβούλιο. το να χαρακτηρίζονται ε, εμπιστευτικά όλα τα έγγραφα εκ των προτέρων δεν είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ε, σοβαρές διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται και κλεισμένων των θύρων, αλλά εδώ δεν συζητάμε αυτό το θέμα. Εδώ Θέλουμε να γνωρίζουμε πώς έχει ψηφίσει το κάθε κράτος μέλος και γιατί. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει στην αύξηση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποφύγουμε το παιχνίδι ε, των ε, αμοιβαίων κατηγοριών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η σκιώδη συζητήτρια των Σοσιαλιστών από την ΠΕΤΗ. Ευχαριστώ. Μιλάω εκ μέρου τη κύρια Ντάρλινγκ, η οποία είναι σκιώδη συζητητριά μα στην Επιτροπή Αναφορών, αλλά και εκ μέρου μου, μια που είμαι συντονίστρια. Ο σκιώδη, η Τζούντι, έχει κάποιε παρατηρήσει να κάνει, γι' αυτό θα σας μεταφέρω στα αγγλικά. Θέλω να ευχαριστήσει και τους δύο συζητητέ για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Πιστεύει ότι η έκθεση καλύπτει όλα τα στοιχεία κλειδί της έκθεσης της Ombudsman και τονίζει ποια είναι η θέση του σώματος απέναντι στα όσα αναφέρει ο Ombudsman. Καταδεικνύονται κίνδυνοι εφόσον δεν αναλυφθεί δράση. Έχοντας ε, δει από πρώτο χέρι στην περιφέρειά της ε, πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η κατάσταση, όταν κάτι πάει στραβά, θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή της έλλειψης διαφάνειας δηλαδή οδήγησε εν μέρη και στο Brexit. Και αυτό το μάθημα πρέπει να το πάρουμε. Γι' αυτό θα πρέπει και το Κοινοβούλιο και όλοι να το συνειδητοποιήσουν αυτό. Κάποιοι έτσι καλλιώς ποτέ δεν θέλουν την αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Πάντως ο καλύτερος τρόπος είναι να ιτηθούν στο δικό τους το παιχνίδι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να λογοδοτούμε όσο γίνεται περισσότερο. Όπω λέει και η Washington Post, η δημοκρατία δεν πρέπει να βρεθεί στο σκοτάδι. Στηρίζει απόλυτα την έκθεση αυτή. Και συνεχίζω στα γαλλικά. Συμφωνώ και εγώ με την Τζούντι και ευχαριστώ και εγώ τους δύο συνεισηγητές. Το έργο τους συνεχίζει το έργο της διαμεσολαβήτριας της κυρίας Ωραίλη. Η έκθεση της Ombudsman βασίζεται στην έρευνά της και δείχνει ότι δεν υπάρχει καθόλου διαφάνεια και υπάρχει και κακοδίκηση. Κάτι το οποίο πλήττει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και τα υπογραμμίζουν όλα αυτά οι συνεισηγητές, ότι η έλλειψη διαφάνειας ε, πλήττει το άνοιγμα, την εγκύτητα στους πολίτες. Συμφωνώ επίσης με την ανάλυση τη Τζούτου Ντάρλινγκ ότι οι χώρες μέλη προσπαθούν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους και να τις φορτώσουν πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρύβονται αντί να λογοδοτούν στους πολίτες. Δεν είναι αυτής της εποχής με τέτοια συμπεριφορά όμως. Οφείλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Εξού και ευχαριστώ για άλλη μια φορά τους συνεισηγητές και τονίζω πόσο σημαντικό είναι το έργο τους αλλά και της κυρίας Ορέλη βεβαίως. Βάσει των διαπιστώσεων και των συστάσεων ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πετύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις ευρωπαϊκές ε, ε, αποφάσεις και να ψηφίζουν ε, ξέροντας ότι θα γίνει γνωστή ψήφος του συγχωρισμένου. Εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη καθυστέρησε το αεροσκάφος. Ε, Άφησα μάλιστα και τη βαλίτσα μου στο αεροδρόμιο και δεν ξέρω πώς ε, θα την ξαναπάρω, αλλά ήρθα. Και σίγουρα θα χρησιμοποιήσω όλο το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου καταρχήν. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λάινεν για την καλή συνεργασία. Δεν ε, συναντιόμαστε συχνά σε αυτόν τον Νίκο, αλλά πιστεύω ότι γίναμε φίλοι βάσει τη έκθεση αυτή. Και θέλω να ευχαριστήσω και τις γραμματείες Πέτη και Αύκο για την προετοιμασία και την υποστήριξη είναι σύντομη η έκθεση, έτσι λοιπόν θα είμαι και εγώ σύντομη. Το κύριο μήνυμα που δίνουμε είναι ότι υποστηρίζουμε τη διαμεσολαβήτρια. Είναι ένα πολύ σημαντικό το θέμα που έχει θίξει. Ο ρόλο των θεσμών, των θεσμικών οργάνων έχει αλλάξει. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτε ε, και θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη η λειτουργία του. Ε, το Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα διαφανέ. Ε, Όλε οι συνεδριάσεις ε, είναι δημόσιες και όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιμα. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια λοιπόν εδώ σε αυτή την αίθουσα. Όμως αυτό φυσικά δεν ισχύει στο Συμβούλιο, δυστυχώς ούτε στις συνεδριάσεις ε, της Κορεπέρ. Όπως ε, δηλώνεται στις συνθήκες, θα πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα έχουν την υποχρέωση να είναι ανοιχτά και διαφανή. Είναι σημαντικό για τη λογοδοσία. Υπάρχει ανισορροπία μεταξύ των συνομοθετών και όταν δεν είναι ικανοποιημένοι οι πολίτε για το αποτέλεσμα, τα κράτη-μέλη μπορούν να καταδείξουν ε, το Κοινοβούλιο και ποιο φταίει, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί οι αποφάσει μα ε, είναι γνωστέ. Όμω αυτό που δεν βλέπει το κοινό συχνά είναι ότι το αποτέλεσμα είναι, ε, προέρχεται από μια διαμάχη μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και συνήθως κατηγορούν τις Βρυξέλλες. Ξέρετε ότι όλα τα καλά πράγματα γίνονται από τις τοπικές κυβερνήσεις και τα κακά πράγματα προέρχονται από τις Βρυξέλλες. Και εμεί ε, τι κάνουμε εδώ, απλώ μετράμε το μέγεθο των αγκουριών. Έτσι λοιπόν, ακόμη και τα Εθνικά Κοινοβουλία ενημερώνονται πάρα πολύ αργά για τις αποφάσει των κυβερνήσεων, αν καν ενημερώνονται. Προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στα σημεία αυτά στην έκθεση τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα, ότι θα πρέπει το Συμβούλιο να ακολουθήσει τις συστάσεις της Ombudsman. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό και να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι εμείς ως Κοινοβούλιο είμαστε υπέρ της διαφάνειας και για μια ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Τόμ. Να περάσουμε ε, στο ECR. Είναι εδώ ο κύριος Σμέτερς, είναι ο κύριο Μαριάς. Όχι, δεν είναι εδώ. Πάμε στο Άλντε. Η Μάιτε, παρακαλώ. Ευχαριστώ και τις δύο Προέδρους. Καταρχήν, ε, ε, ευχαριστούμε τη διαμεσολαβήτρια για το έργο της. Μας φαίνεται εξαιρετική και θέλουμε να την υποστηρίξουμε. Δεύτερον, εγώ πιστεύω ότι υποστηρίζουμε σημείο προς σημείο όλα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Λάινεν, καθώς και από την κυρία Τούμ. Πιστεύω ότι έχουν επικεντρώσει πάρα πολύ καλά τη δουλειά, έχουν κάνει μια πολύ καλή προσέγγιση στην πρόταση ψηφίσματος. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την οδό, οπωσδήποτε. Υπάρχει δυστυχώς μια πολύ διαστραμμένη κουλτούρα από την πλευρά του Συμβουλίου που φτάνει σε καθένα από τα κράτη-μέλη και δρά υπό συνθήκες αδιαφάνειας, δρώντας με έναν τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με την κουλτούρα που ακολουθούμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Παραδείγματο χάρη, όταν ε, ε, γίνεται κατευθυντικό, κατηγορούν τι Βρυξέλλες, όταν αυτοί είναι αυτοί που κυρίω ε, οικοδομούν τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και δεν μπορούν να κρύβονται πίσω ε, από το ρητό «Α, το έκαναν οι Βρυξέλλες». Αυτό είναι πάρα πολύ διαστραμμένο για τη δημοκρατική κουλτούρα και για την ε, δημοκρατική συγκυρία που βιώνουμε στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, όσο εμεί μπορούμε να έχουμε επίπτωση στο έργο αυτό. Θα πρέπει να σκίσουμε πυραιοί για να μην συνεχίσουν να κρύβονται και να απαντήσουν. Είναι καταπληκτική ευκαιρία να γίνει ε, μια συζήτηση για τις συστάσεις αυτές της διαμεσολαβήτριας. Από την άλλη, εμείς θα προσπαθήσουμε, όπως είπε και ο κ. Λένε, να επικεντρωθούμε στα επιμέρους στοιχεία ε, του ψηφίσματος. Δεν θέλουμε να βγούμε εκτός θέματος και σας συγχαίρουμε γιατί είναι ε, πάρα πολύ επικεντρωμένα τα ζητήματα. Θα ήθελα να στείλουμε κάποιες τροπολογίες που αναφέρονται στις διαπραγματεύσεις για το Μητρό Διαφάνειας. Και εμείς έχουμε αρκετά προβλήματα στο να προχωρήσουμε εκεί. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και τη ίδια Μεσολαβήτρια για το έργο της. Ευχαριστώ Μάιτε. Δεν βλέπω την κυρία Σπινέλη για την ΚΟΕ. Και μετά να πάμε στους πρασίνους. Σύμφωνα με τον κατάλογο, η κυρία Κούνεβα επίσης απουσιάζει. Πάμε τώρα στους πρασίνους, η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώ Λάινεν για την σύντομη και σαφή δουλειά που έχει κάνει εδώ. Πρέπει να επιμείνουμε στον πυρήνα, στα κεντρικά θέματα των του δημοκρατικού ελλείμματος της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να φέρονται σαν το Συμβούλιο να είναι διακυβερνητικό σώμα με εμπιστευτικότητα χωρίς κανένα δημοκρατικό έλεγχο. Πολύ βολικό αυτό και πολύ εύκολο να κατηγορεί κανείς άλλους ε, να είναι οι Βρυξέλλες ο αποδιοπομπέος τετράγο όταν τα πράγματα πάμε στραβά. Θα πρέπει επιτέλους ε, το ε, Συμβούλιο να αρχίσει να φέρεται σαν θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συμμετοχή των πολιτών και με διαφάνεια. Χαίρομαι πολύ που βλέπω την έκθεση αυτή, διότι καθιστά απόλυτα σαφές το πρόβλημα όσο τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια δεν μπορούν να παρακολουθούν τι εργασίε ε, και δεν μιλώ μόνο για το πώ ψηφίζει η δική του κυβέρνηση αλλά πώ ε, φέρονται και οι άλλοι Όπω άλλωστε κάνουμε στα κοινοβούλια. Εγώ ήμουν βουλευτή στο Εθνικό Κοινοβούλιο τη Δανία επί πολλά χρόνια. Το Κοινοβούλιο ανακοίνωνε ότι έχουμε αποφασίσει αυτό και αυτό, χωρί να λέει ποιο είπε τι καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία. Αυτό είναι σκανδαλώδε. Και εδώ το Συμβούλιο κάνει ακριβώ αυτό. Θα είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξουμε αυτό, διότι πρόκειται για βαριά ριζωμένες συνήθειες και εργάζονται σαν διπλωμάτες. Εμείς όμως ε, εκλεγόμαστε στις, σε άμεσες εκλογές. Θα πρέπει λοιπόν τις κυβερνήσεις μας αλλά και ε, ο εθνικός τύπος θα πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες. Αυτό βέβαια θα στοιχήσει πολλά, αλλά εάν έχουμε τη διαφάνεια θα μπορεί ο καθένας να παρακολουθεί τι γίνεται εδώ. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και η δική μας έκθεση ζητούν ακριβώς αυτό, να υπάρχει διαφάνεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε οι κυβερνήσει να κατανοήσουν τι διακυβεύεται εδώ πέρα. Το ευρωπαϊκό μέλλον, η αξιοπιστία της Ευρώπης εξαρτώνται από αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαξ Άντερσον. Από τους πράσινους. Θα είμαι σύντομος. Είναι πολύ καλή η έκθεση αυτή. Θα μπορούσαμε να επικρίνουμε ακόμα περισσότερο το Συμβούλιο, αλλά είναι εξαιρετική έκθεση. Πολύ συχνά τόσο σύντομο είναι ο συνάδελφο. like to Να προχωρήσουμε τώρα στο EFTD. Ο Φάμπιο Καστάλτο είναι απόν, ε, δεν τον αντικαθιστά κανεί, αλλά η Ελεονόρα Εύη είναι εδώ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ είμαι στο ίδιο μήκο κύματο, με όσα είπαν ε, οι συνάδελφοι γιατί συμφωνώ απόλυτα. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή για ένα θεμελιώδες ζήτημα. Ένα ζήτημα που χάρη στην Ευρωπαία Δημοσιολαβήτρια και στο έργο που υλοποιεί για να παρακολουθήσει την ε, καλή δίκηση ή μάλλον την κακοδίκηση θα πρέπει να πούμε των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αν ε, δεν ε, ήταν ε, η Ombudsman δεν θα μπορούσαμε να καταγγείλουμε αυτό που σημαίνει εδώ και πολύ καιρό μπροστά στα μάτια μας. Είχα την δυνατότητα, είχαμε τη δυνατότητα να εργαστούμε και στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για την οποία εγώ είμαι η συγγήτρια και την έκθεση που συζητάμε σήμερα την υποδέχομαι πάρα πολύ θετικά γιατί ακριβώς φωτίζει μια προβληματική που εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν έχει επιληθεί. Βλέπουμε μια μεγάλη κριτική απέναντι στο Συμβούλιο, το οποίο συνεχίζει να παραβιάζει τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών λόγω πολύ μικρής διαφάνειας ε, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Συμφωνώ με τις επικρίσεις που έγιναν από τους συναδέλφου, και είναι πράγματι απίστευτο πώς δεν καταγράφονται οι θέσεις των μεμονωμένων κρατών μελών κατά τη διάρκεια τη συζήτηση επί των νομοθετικών φακέλων. Αυτό δεν μπορεί παρά να ζημιώνει τη δημοκρατία και την, ε, να παρεμποδίζει τους πολίτες από την πρόσβαση στα έγγραφα δεν καταγράφονται ε, τα έγγραφα, το δημόσιο μητρό των εγγράφων συνεχίζει να είναι ελιπές, έτσι λοιπόν δεν μπορούν να προσφύγουν εκεί οι πολίτες και επίσης δεν μπορούμε να δεκτούμε και την συστηματική ε, ουσιαστικά ότι τα έγγραφα καθίστανται συστηματικά απόρριτα το κανονισμός του 2001 συνεχίζει να μην έχει αναθεωρηθεί και θα έπρεπε να γίνει αυτό το συντομότερο. Από τη δική μου σκοπιά, Δηλώνω εκ νέου την υποστήριξή μου στην έκθεση αυτή. Θα στείλω και τροπολογίες που θα ενισχύσουν την ανάγκη για μια πλήρη διαφάνεια που επαναλαμβάνω χρειάζεται πλήρης διαφάνεια και πλήρης πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα. Φανώς ό,τι αφορά την νομική, νομοθετική διαδικασία αλλά και τους τριμερείς διαλόγους. Εμείς προς αυτήν την κατεύθυνση εργαστούμε σε αυτή την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Φανέμαντς, για το ΕΝΕΦ, όχι δεν θέλετε το λόγο. Εγώ ελπίζω ότι θα είχατε άλλη άποψη. Όχι ο Ζερόμ Λευλέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Θα ήθελα να συγχαρώ τις δύο εισηγήτριες ε, για το έργο τους. Τα μέτρα που μας προτείνουν, εάν τεθούν σε εφαρμογή, θα έχουμε μια νέα συνταγματική αντίληψη της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που θα μπορούσε να προκύψει. Σε ό,τι με αφορά. Εγώ θα θέσω μία και μόνο τροπολογία. Θα μας επιτρέψει να πάμε κάπως πιο μακριά στο άρθρο 16, παραγραφος 1, όπου ζητάμε συστηματικά να καταγράφεται η ταυτότητα των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν καλό να καταγράφουμε συστηματικά την ε, ταυτότητα των κυβερνήσεων και των αντιπροσώπων. Γιατί σε κάποιες χώρες γίνεται ένα παιχνιδάκι και συνήθω το εξή, να λένε Α, δεν έχουμε ψηφίσει επίσημα, αλλά δεν, επομένω δεν είμαστε υπεύθυνοι. Όμω, ε, στη σπάνια περίπτωση που έχουμε ψηφοφορία, θα λένε κάποιοι, Α, εγώ δεν ήμουν εκεί. Ακόμη και οι υφυπουργοί ε, για ε, σε ευρωπαϊκές υποθέσεις. Αναφέρομαι ε, σε κάποιο από τη χώρα μου, παραδείγματος χάρη, όταν δεν είναι πλέον Υφυπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και έχουν αναλάβει, παραδείγματος χάρη, άλλα καθήκοντα, είναι πρόεδροι παραδείγματο χάρη των κομμάτων σε προκλητική περίοδο, αρνούνται το τι συνέβη. Ε, και αυτό επιτρέπει σε κάθε δημαγωγό να πει οτιδήποτε κάποιο μήνε ή κάποια χρόνια πριν, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Έτσι λοιπόν, ε, θέλω να επισημάνω ότι το σύνολο των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάθε φορά που είμαστε παρόντε σε μια αίθουσα, είναι δημόσιο αυτό. Όταν απουσιάζουμε, επίση είναι δημόσιο. Και κάθε φορά που ψηφίζουμε, όποια και αν είναι η δική μα ψήφο, είναι κάτι δημόσιο. Και όταν λείπουμε, πάλι αυτό είναι δημόσιο. Έτσι λοιπόν, ε, σε 10-15 χρόνια κάποιο μπορεί να ξέρει τι ψήφισα, αν ήμουν εκεί, αν έλειπα και αναλαμβάνω τι ευθύνε μου και ακόμη ε, και ο καθένα σε μια προεκλογική εκστρατεία είναι ελεύθερο να ψηφίσει ότι θέλει, υπάρχει ένα φόβο τη ευθύνη. Νομίζω ότι αυτή η αρχή θα πρέπει να ισχύει και για τα μέλη των κυβερνήσεων. Και ε, πέρα από μια πρόταση κειμένου για τη διαφάνεια, νομίζω ότι κυρίω αφορά μια πρόταση για την καταπολέμηση της υποκρισίας. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ζερόμ. Ο Έλματ Πρόκ είναι ο τελευταίος που έχω στον κατάλογό μου, σκιώδης εκ μέρου του ΕΛΚ. Κυρία Πρόεδρε, ε, Πράγματι πρόκειται για υποκρισία. Ένα από τα σημαντικά προβλήματά μας είναι ότι οι κυβερνήσεις όταν συμφωνούν με κάτι στο ε, συμβούλιο, το οποίο δεν είναι πολύ δημοφιλές στην πατρίδα, τους κάνουν σαν να μην ήταν εκεί. Το θέμα αυτό είναι ένα από τα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που έχουμε. αναφέρθηκαν και οι ψευδείς ειδήσει και αυτό δυστυχώς είναι αλήθεια. Να το πω ως εξής. Συμφωνώ με την πρόθεση της έκθεσης αυτής. Συμφωνώ και με την έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. Ε, πρέπει να πετύχουμε περισσότερη διαφάνεια ακριβώς για τους λόγους που περιγράφονται. Αλλά όσον αφορά την μέθοδο έχω κάποιες παρατηρήσεις. Λέμε ότι θα πρέπει να είναι όλα ε, διαφανή και ανοιχτά ε, στο Συμβούλιο. Αλλά ας δούμε εμείς τι κάνουμε. Ε, η διάσκεψη των Προέδρων συνεδριάζει δημόσια, οι πολιτικές ομάδες συνεδριάζουν δημόσια. Όχι. Θα πρέπει λοιπόν ε, να περιμένουμε και εκείνοι να κάνουν ε, διάφορες διακρίσεις, αλλά και αυτό είναι υποκρισία. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε μήπως προβάλλουμε επιχειρήματα τα οποία θα μπορέσουν να στρέψουν εναντίον μας μετά. Ζητάμε κάτι το οποίο στην ε, συνταγματική συνέλευση καταψήφισαν ε, τα μέλη της μέσα στο πρώτο μισάωρο. Το Συμβούλιο Υπουργών, το Συμβούλιο Υπουργών να ε, συνεδριάζει πάντα δημόσια. Αυτό ήταν το σημείο εκκίνησης. Άλλωστε, μετά από τη συνταγματική συνέλευση είχαμε μόνο ένα Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά άλλωστε αυτό θα πρέπει να ισχύει όταν νομοθετεί το Συμβούλιο. Το, Υπουργείο, το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικού, ε, Εξωτερικών ε, δεν νομοθετεί, οπότε και εκεί δεν θα πρέπει να ισχύει αυτό. Μιλάμε εδώ για τις περιπτώσεις όπου ενεργεί ως νομοθέτης το Συμβούλιο. Σημαντικό είναι λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο να συνεδριάζει σε κοινοβουλευτικό πλαίσιο και κάθε κυβέρνηση ε, να ε, ψηφίζει ανοιχτά, να γνωρίζει ο πολίτης τι ψηφίζει η κάθε κυβέρνηση. Και από εκεί και μετά μπορούμε να εξετάσουμε τα επόμενα βήματα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα λειτουργούσε μόνο εάν τα επιμέρους υπουργικά συμβούλια δεν ε, έχουν πια ε, νομοθετικές εξουσίες. Έτσι όλα θα περνούν ως σημεία άλφα. Τα επιμέρους υπουργικά συμβούλια θα πρέπει να είναι οι επιτροπές του ε, ενιαίου Υπουργικού Συμβουλίου. Και με αυτή τη βάση θα έχουν κοινοβουλευτική δομή και κατόπιν θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε ε, ποιοι τομείς θα είναι δημόσιοι και ποιοι όχι. Αυτή τη στιγμή που ε, το Υπουργικό Συμβούλιο λειτουργεί ως άνω βουλή, ως δεύτερη βουλή, θα πρέπει να έχει ακριβώς ε, αυτή τη δομή. Ας εξετάσουμε λοιπόν μήπως μπορούμε να οργανώσουμε τη δομή ώστε να μην μπορούν να στρέψουν εναντίον μας τα επιχειρήματά μας και να εργαστούμε με βάση τα αποτελέσματα της ε, συνταγματικής συνέλευσης. Η συνάδελφος Σεμπρέσο είχε εργαστεί πάνω στο θέμα αυτό. Και το κατά πόσο θα πρέπει να είναι όλα δημόσια, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά ε, τις συνεδριάσεις που δεν διενεργούμε εμείς σε δημόσια δεν μπορούμε να ζητάμε το Συμβούλιο ε, να τις ε, δημοσιεύει. Επίσης, ε, και τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν πλεονεκτήματα από αυτό. Κάθε κράτος μέλος έχει το δικό του τρόπο να ελέγχει την κυβέρνησή του, να ελέγχει τη συμπεριφορά του στο Συμβούλιο. Οι κυβερνήσει υπαγορεύουν την συμπεριφορά εντό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα πρέπει να φροντίσουμε ε, τα κοινοβούλια των κρατών μελών να μπορούν να ελέγχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις κυβερνήσεις τους. Ε, το Συμβούλιο στο σύνολό του όμως δεν πρέπει να το ελέγχουν τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά εμείς. Αυτό είναι δικό μας καθήκον. Ε, τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων θα πρέπει να ελέγχουν τη συμπεριφορά του δικού τους αντιπροσώπου στο Συμβούλιο, όχι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο σύνολό του. Ευχαριστώ. Εποφελούμε από αυτή την ευκαιρία να μιλήσω ως πλευροβουλευτής, γιατί το βρίσκω απαράδεκτο όταν κοιτάω την παρουσία του Συμβουλίου. Θέλω να σας στείλω ένα μήνυμα. Σημειώνετε λοιπόν. Μέχρι αυτή τη στιγμή η Προεδρία, η Αυστριακή του Συμβουλίου δεν ε, προχώρησε στην ε, δέσμευση που είχε αναλάβει ο Προεδρεύων στις 11 ε, Ιουλίου όταν είχε πει ότι δεσμεύεται να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο του Συμβουλίου όσον αφορά τον ε, συνεχιζόμενο προβληματισμό για τους κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν την νομοθετική διαφάνεια. Αυτό τον Ιούλιο. Τώρα είμαστε τέλη Σεπτεμβρίου και τίποτα δεν πήραμε από το Συμβούλιο. Βρίσκω ότι είναι απαράδεκτο αυτό. Και εδώ δεν μιλάω σαν πρόεδρο μια κοινοβουλευτική επιτροπή, η Δανούτα προεδρεύει. Εγώ μιλάω σαν απλή ευρωβουλευτή. Επίση, ο κύριο Λάινεν λέει στο Συμβούλιο: Σταματήστε να εργάζεστε σαν διπλωματικό σώμα, αλλά εργαστείτε σαν κοινοβουλευτικό δημοκρατικό σώμα. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς εσάς. Η... Κύριε Χούμπνερ, ευχαριστούμε Σεσίλια, δεν ξέρω αν οι δύο συνεισηγητέ θέλουν πάλι το λόγο πριν κλείσουμε. Ε, Γιάννα πρώτα ή εσείς. Γιάννα Τόμ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για την ε, βοήθειά σας, για τις παρεμβάσεις σας. Εμένα με βοήθησαν πραγματικά πολύ, ιδιαίτερα αυτά που είπε ο κύριος Μπροκ, ο οποίος εδώ και χρόνια τα έχει ξαναπεί και δεν έγινε τίποτα στο Συμβούλιο. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά η προσέγγιση μας ε, θα ακολουθήσει ένα διαφορετικό πρίσμα, θα βρούμε ένα διαφορετικό δρόμο για να πετύχουμε το στόχο μας αυτή τη φορά. Και πράγματι είναι θλιβερό που το Συμβούλιο δεν, δεν απάντησε ούτε στην επιστολή της Ομπουτσμεν, ούτε τίποτα. Και είναι εδώ και σιωπούν. Εγώ μίλησα με διάφορους εκεί και είπα ότι δεν είναι διπλωματία ε, που χρειάζεται. Η αντιμετώπιση τους πραγματικά ήταν δυσάρεστη. Ο κύριος Λάιναν. Ναι, πολύ σωστά είχε πει συνάδελφος ότι ε, η διαφάνεια στο Συμβούλιο θα επιτρέψει μια νέα συνταγματική αντίληψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δείξει ότι το Συμβούλιο είναι νομοθέτης και όχι ε, ένα διακυβερνητικό σώμα. Η διαφάνεια όσον αφορά τις θέσεις των ε, κρατών μελών σημαίνει ότι δεν θα θεωρείται πια ότι οι Βρυξέλλες είναι μια ξένη δύναμη με την οποία δεν έχουν καμία σχέση τα κράτη-μέλη. περισσότερη διαφάνεια ε, θα απέτρεπε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ο σοφός Έλμαρ Μπρόκ παρόλα αυτά έχει άδικο, διότι η Κορεπέρ αντικατοπτρίζει αντιστοιχεί στις δικές μας επιτροπές και το ε, Συμβούλιο ε, αντιστοιχεί στη δική μας Ολομέλεια. Θα πρέπει λοιπόν ε, να συνεδριάζουν δημόσια. Δεν ε, θέλουμε να δημοσιεύουμε τα εμπιστευτικά έγγραφα της ε, κάθε αντιπροσωπείας, όπως άλλωστε δεν δημοσιεύουμε και εμείς όλα τα δικά μας έγγραφα. Στο σημείο 14 λέμε άλλωστε και εμείς ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να, θεωρεί, να θεωρείται νομοθετικό σώμα Και το να υπάρχουν 16 Υπουργικά Συμβούλια δεν προβλεπόταν αρχικά. Ε, δείχνει όμως ε, το πόσο ε, έχει διευρυνθεί το σύστημα. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις σας και περιμένουμε τις τροπολογίες σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται αυτή η κοινή συνάντηση. Την τελική ψηφοφορία θα την κάνουμε 21 Νοεμβρίου. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 3η Οκτωβρίου, μέχρι τη λήξη των εργασιών την ημέρα εκείνη. 3 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος των εργασιών. Ευχαριστώ πολύ. Και η ΑΦΚΟ πρέπει να πάει σε άλλη αίθουσα για τη δικιά μας συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σεσίλια, που μας έδωσε αυτή την